Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της μερισίας διατάξεως, δηλαδή την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων. Αγαπητοί συνάδελφοι, εφέτος είναι το έτος των συνεταιρισμών, το οποίο εορτάζουμε, που είναι ε, μέρος της αλληλέγγυας οικονομίας και έχουν σημαντικό σημαντικό ρόλο για την οικονομία και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, ε, εφόσον πάνω από 160 εκατομμύρια επιχειρήσεις εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά μέλη αυτών των επιχειρήσεων και 4,5 εκατομμύρια συνεργάτες πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα καλά εδρεωμένο σύστημα έχει αποδειχθεί στο παρελθόν σταθερό και ε, υλοποιεί και συμβάλλει στην πρόθεση των σόχων του 2020 όχι από πλευράς μόνο κοινωνικής απασχόλησης αλλά και όσον αφορά το, ε, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόθεση της κοινωνίας. Γι' αυτό και πρέπει να αξιολογήσουμε την σημασία των συνεταιρισμών και να την αξιοποιήσουμε. Έχω την ε, Έλλην Ρέγνερ, σκιώδη συγγήτρια την οποία ευχαριστώ που κάθεται ακόμη έτσι αργά σήμερα και θέσαμε το ερώτημα πώς το καταστατικό των συνεταιριστικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να τροποποιηθεί διότι με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Δικαίου ε, μειώθηκε η ε, σημασία του θεσμού αυτού και μόνο 17 ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες έχουν δημιουργηθεί με λίγους ε, εργαζομένους πράγμα το οποίο οφείλεται στο πολύ πολύπλοκο καταστατικό το οποίο ε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ε, διασυνοριακό έργο και γι' αυτό πρέπει να επεξεργαστούν και το καταστατικό, να μην μειώσουμε τις προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε, αλλά εφόσον από πλευράς απασχολήσεως δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την εξέλιξη, θα πρέπει να υπάρχει μία πρόθεση της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας και θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα του τομέα αυτού είναι πολύ κατακαιρματισμένες παρά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ε, επαρκές ε, προσωπικό που να ασχολείται με τον τομέα αυτό και ε, ούτως ή άλλως διανύμεται σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας και να μπορέσει να υπάρχει μία διαδικασία για μη συστηματική παραβολή των των διαφόρων συστημάτων που ισχύουν στον τομέα των συνεταιρισμών και των ε, ε, αλληλεγγύων ε, εταιριών κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις 12 δράσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί ε, των οποίων μόνο τρεις έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής δηλαδή δεν υπάρχει ένα εκτενές επιμορφωτικό πρόγραμμα και μία αναγνώριση των ιδιομορφιών των συνεταιρισμών θα θέλαμε επίσης οι συνεταιρισμοί στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών και ε, της ρυθμίσεως να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν είναι δυνατόν οι τομείς οι οποίοι ε, προωθούνται να χρειαστεί ε, να αλλάξουν μετά την κρίση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει για να στηρίξει την συνεταιριστική βιομηχανία. Ευχαριστώ. Έχουμε την, ε, πέντε συναδέλφους που ζητούν το λόγο, εκ των οποίων ο πρώτος είναι ο κύριος Μικολάσεκ. Η αποτελεσματική λειτουργία και η συμμετοχή των εργαζόμενων είναι κάτι το σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι ευρωπαϊκές εταιριστικές εταιρείες προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών τους αλλά συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προωθώντας καινοτομίες την παροχή ε, εφοδίων σε, τόσο σε αγροτικές όσο και αστικές περιοχές υπάρχουν πάνω από 160.000 συνεταιρισμοί που παρέχουν απασχόληση σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες και είναι λυπηρό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο 17 ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες έχουν συσταθεί μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει, δυστυχώς έλεξε ο χρόνος μου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Νταντσίλα τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Η χρηματοοικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε πλήττει και τις συνεταιριστικές εταιρείες. Συνεταιριστικές εταιρείες, με συγχωρείτε. Ε, που δημιουργούν εργασία σε τοπικό επίπεδο και δεν μπορούν να μετεκατασταθούν. Δίνουν εργασία και σε πολλές γυναίκες. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν πολύ περισσότερο τέτοιες πρωτοβουλίες, ακόμα και σε χώρες όπου οι συνεταιρισμοί αυτοί δεν έχουν τον ιστορικό χαρακτήρα που διαθέτουν άλλες. Τουλάχιστον έτσι ώστε να μην διατρέχουν τον κίνδυνο να, μετε... να εγκατασταθούν αλλού. Έχει μεγάλη σημασία για την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαμπασούμπορ ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση του συναδέλφου Γκίγκολτ σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών σε σχέση με τη συμμετοχή των ευρωπαίων εργαζομένων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό διότι στη χώρα μου, στη Ρουμανία όπως και σε άλλα κράτη-μέλη ο θεσμός των συνεταιρισμών είχε ε, μειονεκτήσει πάρα πολύ κατά την κομμουνιστική εποχή και από το 2010 οι εξελίξεις δεν έχουν αποσαφινιστεί. Υπάρχουν υπερβολές. Χρειάζεται λοιπόν μία πιο ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στους συνεταιρισμούς και λυπούμε ότι πρόκειται για μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ρεγκιάνοβα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεταιρισμοί στην Ευρώπη που απασχολούν 4,7 εκατομμύρια εργαζόμενους και μόνο, δεν είναι μόνο οι μέτοχοι σημαντικοί αλλά και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείε. Πρέπει να, να λάβουμε υπόψη τη σημασία αυτών των εταιριών για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία υπάρχει το καθεστώς, το καταστατικό το οποίο είναι το κοινό εργαλείο στην Ευρώπη αλλά οι συνεταιρισμοί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού μοντέλου. Χρειάζονται λοιπόν την υποστήριξή μας αξίζουν την υποστήριξή μας και το κείμενο αυτό θα πρέπει να εστιαστεί στις ειδικέ ανάγκες των υπαλλήλων και των εργαζόμενων σε αυτές ε, τις ε, συνεταιριστικές εταιρείες. Ήταν καλό εάν μπορούν να γίνουν συνειδιοκτήτες οι εργαζόμενοι των ε, συνεταιριστικών αυτών εταιριών. Ευχαριστώ. Η Εύελιν Ρέγνερ τώρα είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα από την αρχή να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γκίγκολτ διότι ε, και ε, σαν ε, ε σκιώδη με ενέπλεξε άμεσα στην διαδικασία και όπως ανέφερε υπάρχουν 17 μόνο ευρωπαϊκά ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί και φέτος που είναι το, έτρο, το έτος των συνεταιρισμών δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν βλέπουμε μία θετική εξέλιξη. Σε τι οφείλεται αυτό. Αφενός είναι οι διατάξεις οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες και ίσως ε, δεν χρειάζεται να υπάρχει μία τέτοια διασυνοριακή συνεργασία. Προσπαθούμε ε, με τα ε, διάφορα μέσα να βοηθήσουμε τους συνεταιρισμούς να αναβιωθούν και ξέρω ότι έχω μόνο ένα λεπτό αλλά θα ήθελα τελειώνοντας να τονίσω τη σημαντική σημασία της εκθέσεως αυτής η οποία θα πρέπει και στο μέλλον να ε, διεκπαιρεωθεί πολύ προσεκτικά. Σας ευχαριστώ και τώρα θέλω να παρακαλώ καλέσω την ε, Επίτροπο Βασιλείου να μας παρουσιάσει την άποψή της. Ο χαιρετίζει το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Το 2012 είναι το Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Αναφέρεται σε μια ουσιαστική συμβολή στην αναθεώρηση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας. Λέει ότι μπορεί να, να προβάλλει την αναγνωρισιμότητα και να τονίσει το θετικό ρόλο που το ε, συνεταιριστικό εργασιακό πρότυπο μπορεί να συμβάλλει στους στόχους του 2020. Έχει παραμεληθεί ο ρόλος των συνεταιρισμών για κάποιο διάστημα μέχρι τη στιγμή που ο κόσμος άρχισε να βιώνει την, ε, οικονομική κρίση, το ενδιαφέρον στην ικανότητα των συνεταιρισμών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ευμάρεια αυξάνεται και πάλι. Είναι γεγονός ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις που τηρούν τις συνεταιριστικές αξίες μπόρεσαν να αντισταθούν στις επιπτώσεις της οικονομικής και, χρηματο, και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η έκθεση αναφέρεται στις σκέψεις της Επιτροπής για το μέλλον του εταιρικού δικαίου σε συνδυασμό, σε συνδυασμό με την επιχειρηματιστική πρωτοβουλία που υιοθέτησε πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή σημειώνει ειδικότερα την πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του καταστήματος της Ευρωπαϊκής Εταιριστικής Εταιρείας, η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή την εταιρεία, η ενίσχυση των συνεταιρισμών και η παροχή ιδιαίτερης προσοχής στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Θέλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Γκίγκολ και τα εκπροσώπους της Επιτροπής Γυναικών για τη συμβολή του. Η Επιτροπή διαπίστωσε, όπως αναφέρεται άλλωστε στην έκθεση, ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τα μέσα που έχει δημιουργήσει ο κανονισμός. Μόνο 24 ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν από το 2006, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού. Στις 23 Φεβρουαρίου 2012 η Επιτροπή ενέκρινε μία έκθεση για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού την οποία έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα. Το κείμενο αποκαλύπτει ότι το μέσο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και αυτό είναι εμπόδιο στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Κανονισμού. Γι' αυτό η Επιτροπή θα οργανώσει δύο μεγάλες διασκέψεις για να, έρθει, να διαβουλευθεί με τους, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς μπορεί να πλουστευτεί το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρεία. Η μία διάσκεψη θα γίνει τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες με συμμετοχή επιτρόπων Καγιάννη και Μπαρνιέ <coughs> και οι άλλοι στην Κύπρο στη διάρκεια της ε, Κυπριακής Προεδρίας το Σεπτέμβριο. Η Επιτροπή σκοπεύει να επανέλθει στο Κοινοβούλιο αφού θα έχετε εξετάσει την έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία των, διαβουλε... των διαβουλεύσεων με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές στη διάρκεια των δύο αυτών διασκέψεων. Η ανάλυση των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης για την απλούστευση της νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Σταθεριστική Εταιρεία θα επιτρέψει ε, θα επιτρέψει επίσης την προώθηση του ευρωπαϊκού δικαίου και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Έκλεισε η συζήτηση. Αύριο στις 12.30 θα υπάρξει ψηφοφορία και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο θέμα της σημερινής